Λοιπόν, περνάμε τώρα στι επεξηγήσει ψήφου. Πρώτα στην έκθεση Φλάσακ, περιφερική πολιτική ω τμήμα των ευρύτερων κρατικών επιδοτήσεων και των κανονισμών για αυτού. Ε, πρώτη, η συνάδελφο Μπαράτσιου.